Θα περάσουμε αμέσως στο σημείο 27, όπως είχαμε αποφασίσει χθε. Είναι η γνωμοδότηση της κυρίας Κίνγκα Γκέντς προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας για το κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Δημιουργική Ευρώπη. Έχετε το λόγο, κυρία εισηγήτρια, για να μας παρουσιάσετε την γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Στα γρήγορα, θα ξεκινήσω λοιπόν. Γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα αυτό, η Δημιουργική Ευρώπη, είναι ο διάδοχος των προηγουμένων προγραμμάτων, όπως έγινε και σε άλλους τομείς, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, συνδυάζονται διάφορα προγράμματα μεταξύ των. Μία εκ των ανησυχιών μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα ετήσια προγράμματα εργασίας θα αντικατοπτρίζουν όλους τους ε, στόχους, σε αυτή την περίπτωση το Media, το Media Mondus και τα προηγούμενα πολιτιστικά προγράμματα. Υπάρχουν κάποια μικρομερίδια τα οποία καθορίζονται ε, εντός του προγράμματος και ο στόχος και ο βασικός ο αντικειμενικός σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να διασφαλίσουμε ότι θα καλύπτονται όλες οι πηγές της πολιτιστικής βιομηχανίας, οι οποίες θα δημιουργήσουν και θέσεις απασχόλησης. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι, καθώς γνωμοδοτούμε, να επικεντρωθούμε στις κοινωνικές πτυχές και στις κοινωνικές ευαισθησίες στον τομέα αυτό. Αφενός αυτό που θα θέλαμε ε, να καταθέσουμε ως τροπολογία είναι μια τροπολογία που θα περιλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο τα πολιτιστικά δικαιώματα και τις ευάλωτες ομάδες, ε, μειονότητες και ούτω καθεξής, να μπορούν δηλαδή και αυτές οι ομάδες ε, να διεκδικούν τα πολιτιστικά τους δικαιώματα και ε, να μπορεί αυτό να περάσει και στους πολιτιστικούς οργανισμούς και αυτό θα θέλαμε να αντανακλάτε όχι μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις διότι γνωρίζουμε ότι ε, υποεκπροσωπούνται αυτές οι μικρές επιχειρήσεις όταν αναφερόμαστε σε τέτοια μέσα. Θα θέλαμε επίσης ε, να εμπλακούν περισσότερο και οι νέοι και να λάβουν περισσότερη υποστήριξη ε, και μικροχρηματοδότηση σε περίπτωση που απαιτείται και επίσης θα θέλαμε να υπάρχει και μια γεωγραφική ισορροπία και να λάβουμε υπόψη και τις περιοχές που υπάρχει μικρότερη δυνατότητα παραγωγής και μικρότερη αγοραστική δύναμη και να ε, συμπεριληφθούν λίγο καλύτερα σε αυτές τις ε, διασυνοριακές ανταλλαγές. Και σε γενικέ γραμμέ νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού τομέα και θα πρέπει να υπάρχουν και στεναροί δείκτε που θα αποδεικνύουν τι ακριβώ συνέβη, πώς δαπανούνται τα κονδύλια και πώ μπορούμε να εξελίξουμε το ετήσιο πρόγραμμα για τι επόμενε χρονιέ. αντλώντα διδάγματα από τα όσα ξέρουμε και να γίνεται και λίγο νωρίτερα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λίγα πράγματα και για το χρονοδιάγραμμα να σα πω. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 14 Ιουνίου, εξέταση των τροπολογιών στι 10 Ιουλίου και ψηφίζουμε στις 19 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος το λόγο. Η κυρία Χίρς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, τη συντάκτρια της νομοδότησης καταρχάς. Νομίζω ότι έχετε συμπεριλάβει μια πολύ σημαντική πτυχή εδώ. Το θέμα των μειονοτήτων ε, και της ε, πιο ευάλωτες ομάδες. κάτι το οποίο είχαμε παραβλέψει λίγο στο παρελθόν. Θεωρώ λοιπόν θετικό το γεγονός ότι γίνεται μία σε αυτό και ελπίζω να ενισχύσει την ε, προοπτική της απασχόλησης η προσθήκη αυτή. Νομίζω ότι είχαμε πολύ καλές ιδέες που έχουμε ακούσει και εμείς θα θέσουμε ως μέσα τροπολογίες και ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία. Ε, So if you withdraw, there's no more uh, on my... δεν έχω καθόλου στο... Δεν έχω κανέναν άλλο στον καταλογό μου, αν δεν θέλετε εσείς να μιλήσετε. Η Κομισιόν έχει κάποιον εκπρόσωπο εδώ. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Τα σημειώνουμε. Τρία στοιχεία. Για τις ε, πιο ευάλωτες ομάδες και τις κοινωνικές πτυχές, ε, να σας πω ότι ένα σημαντικό στοιχείο στην δημιουργική Ευρώπη είναι η ανάπτυξη οπτικοακουστικών ε, πτυχών και μας ενδιαφέρουν και κοινωνικές πτυχές και ένα από αυτά είναι να προσεγγίσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι σημαντικό αυτό ε, έχετε δίκιο, αλλά ήθελα να διευκρινίσω ότι το κοινωνικό σκέλος είναι κάτι το οποίο ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε αυτό το ακουστικό κομμάτι του προγράμματος. Επίσης, μας ενδιαφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι οργανώσεις περιλαμβάνονται στον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και υπάρχει σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2003 που ορίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον ορισμό περιλαμβάνονται και οι, μικρο, οι πολύ μικρής ε, κλίμακες επιχειρήσεις. Να σας πω επίσης ότι εμείς συμφωνούμε και θεωρούμε ότι συμπεριλαμβάνονται γιατί συμπεριλαμβάνονται στον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μια τρίτη διευκρίνηση, συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν δείκτες ε, προκειμένου να αξιολογήσουμε ότι ε, ήταν καλή η απόδοση του προγράμματος και είχε σημαντική επιρροή και αυτό σκοπεύουμε να το κάνουμε ούτως ή άλλως σε όλα μας τα προγράμματα. Σε όλα τα προγράμματα έχουμε συμπεριλάβει δείκτες για τους πιο γενικούς αλλά και τους πιο συγκεκριμένους στόχους που όπως τους αποκαλούμε πρέπει να είναι ευφυείς, δηλαδή να είναι συγκεκριμένοι, να είναι μετρήσιμοι και να μπορούμε να τους επιτύχουμε συν το χρόνο είναι περιορισμένος ο αριθμός των δεκτών που υπάρχουν στη νομική βάση για τους γενικούς και συγκεκριμένους στόχους, αλλά ε, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε και άλλους δείκτες ε, για να βλέπουμε την απόδοση του προγράμματος και σκοπεύουμε να μετρήσουμε και τις ποιοτικέ πτυχές και όχι μόνο τις ποσοτικές πτυχές. Η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, η οποία αναφέρεται στη νομική βάση, είναι ένα εκ των μέσων ε, το οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να δούμε και τις ποιοτικέ πτυχές. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει άλλος, εισηγητρία. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, όχι εγώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ουγγρικά. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για αυτή την έκθεση πρωτοβουλία για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, αν και τα περισσότερα στον τομέα αυτών ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, έχει σημασία να έχουμε μια παρουσία στο θέμα. Ζούμε μια κρίση διαρκείας στον πολιτισμό, στην παιδεία, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου και ούτω καθεξής. Προσπαθούμε επίσης να συγκεράσουμε προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας για να μην χάσουμε μια ολόκληρη γενεά. Τα κράτη μας, οι χώρες μας, αντιμετωπίζουν σοβαρότερες προκλήσεις, προσπαθώντας να εξορροπήσουν την αγορά εργασίας. Άνθρωποι με σημαντικά προσόντα, συνήθως ακόμη βρίσκουν δουλειά, αλλά στην περίπτωση υπερπροσφοράς και εκεί θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Χρειάζεται περισσότερη λοιπόν επαγγελματική εκπαίδευση για εργατικό, δυναμικό, για τεχνίτες, για να διονύσουμε και μερικές παραδόσεις. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη της το περιβάλλον. Επιτρέψτε μου να ευστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη να προσαρμοστούμε σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι νέες γενιές βεβαίως θα το βρουν πιο εύκολο να αντιμετωπίσουν δηλαδή τι σύγχρονε προκλήσεις. Αυτά και είμαι στη διαθεσία για να συζητήσουμε τι τροπολογίε. Ευχαριστώ. Η συγχυτρία. Με συγχωρείτε για την παρεξήγηση. Έχω δύο λόγια να πω. Ναι. Καταρχήν χαίρομαι που το σχέδιο κειμένου της Κομισιόν μιλάει για την ανάπτυξη ακροατηρίου, όπως λέμε. Είναι μια περιεκτική γενική προσέγγιση, αλλά έχει μεγάλη σημασία να δώσουμε ευκαιρίες και σε ευπαθείς ομάδες, σε μειονότητες, μεταξύ άλλων, διότι είναι φορείς κουλτούρας. Συνεπώς, ε, συμφωνώ με την πρόταση αυτή, αλλά πρέπει να διευρυνθεί. Επίσης, για τις ε, νέες επιχειρήσεις ε, που τώρα ξεκινούν, έχει μεγάλη σημασία να εξασφαλίσουμε μικροχρηματοδοτήσεις για να ξεκινήσουν αυτές οι επιχειρήσεις να λειτουργούν και να υποστηρίξουν και άλλους τομείς της οικονομίας. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα. Άκουσα επίση για δείκτε, ότι αναπτύσσετε νέου δείκτε για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων και για να θέσουμε στόχους για του χρόνου. Σημαντικό. Αλλά πρέπει να διαβάσουμε προσεκτικά και την ανάλυση επιπτώσεων με βάση αυτού τους δείκτε, για να δούμε πού πήγαν, πού μας πήγαν οι αποφάσει οι δικέ μα και της Κομισιόν. Έχουμε 7 χρόνια πίσω μας που μας δίνει την ευκαιρία να σταθμίσουμε ακρίβεια τι πετύχαμε. Πρόεδρος, όπως είπε η συγγήτρια, ...14 Ιουνίου 12 το μεσημέρι προθεσμία κατάθεση πολιγιών, 10 Ιουλίου έχουμε τη σύντηση και η ψηφοφορία την ίδια μέρα 19 Σεπτεμβρίου. Και δίνω το λόγο στον κύριο Μπέκερ για να μας μιλήσει για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ή την πρόθεση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας. Έκθεση πρωτοβουλίας, κύριε Ισηγητά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Χαίρομαι πάρα πολύ που η παρθενική μου έκθεση αφορά το οικοσύστημα του επιχειρήν. Σας λέει πάρα πολλά ο τίτλος ήδη για τη στοχοθεσία, το να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα για την προώθηση του κοινωνικού επιχειρήν ως κομβικού δράστη στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας. Ο στόχος είναι να φανεί το πνεύμα <clears throat> της έκθεσης αυτής που ελπίζω ότι θα συναντήσει θετική ανταπόκριση από τους συναδέλφους και καλή συνεργασία. Η κύρια ενασχόληση της έκθεσής μου είναι η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας ώστε να δημιουργήσουμε τις βάσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της καινοτομίας και του επιχειρήν. Αυτό βέβαια το θέμα συνδέεται με πολλές άλλες πτυχές της κοινωνικής οικονομίας, ε, συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την, και το Κοινωνικό Επιχειρήν, το πρόγραμμα για την μεταλλαγή και την καινοτομία και συνδέεται και με την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Βέβαια υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ των δύο ζητημάτων και έχει όμως παρόλα αυτά κάποια επαφή με το θέμα που μας απασχολεί. Θα ήθελα λοιπόν να έχω τη συνεργασία των συναδέλφων για να διαμορφώσω καλύτερα την κατευθύνουσα φιλοσοφία αυτής της έκθεσης. Γιατί εγώ από τη δική μου πλευρά θεωρώ ότι είναι μεγάλη σημασία πέραν των κανόνων και των βασικών προϋποθέσεων να δημιουργήσουμε <clears throat> επαρκές έδαφος για μια φάση που δεν υπήρξε ποτέ στην ε, έννοια του κοινωνικά επιχειρήν, μια φάση που θα επιτρέψει τη δημιουργία καινοτομίας και θα εμπλέξει ιδίως τους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις ελπίδες για μια πράσινη και λευκή μορφή του επιχειρήν. Ελπίζουμε λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να περάσουμε μια φάση δοκιμασίας και πειραματισμού και θα επιτύχουμε τη συμμετοχή και την εμπλοκή των νέων ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλο αυτό το δυναμικό που υπάρχει. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους συνεργάτες μου, θέλω να ευχαριστήσω και την γραμματεία της Επιτροπής, μου, της Επιτροπής μας και την γραμματεία της πολιτικής μου ομάδας που με βοήθησε ιδιαίτερα. Δεν έχω να πω τίποτα για τις ε, προθεσμίες, γιατί ξέρω τα λέει καλύτερα η πρόεδρος μας και της αφήνω αυτό το έργο. Απλώς θέλω να τονίσω ότι πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε μια σημαντική συνεισφορά στην κοινωνική οικονομία μαζί με όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Κίγκαγκόντ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι σκιώδη εισηγήτρια από πλευρά σοσιαλιστών και θα ήθελα και εγώ να σας πω τις απόψεις μου. Συμφωνώ πολύ με τον εισηγητή, τον κύριο Μπέκερ, ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Εν καιρό κρίσης δε ακόμα πιο σημαντική για να υπάρχουν θέσει εργασία ε, και στο κοινωνικό τομέα σε αυτές τις γυράσκουσες κοινωνίες όπου ο τομέας της υγείας ε, και της ασφάλειας γίνεται όλο και πιο σημαντικός και είναι καλό να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εναρμονίσουμε και το χρηματοδοτικό αλλά και το νομικό ε, περιβάλλον για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Θα ήθελα να επικεντρώσουμε το σχέδιο κειμένου μας λίγο καλύτερα στους ορισμούς, διότι υπήρχαν ορισμοί στο παρελθόν και καλό θα ήταν να ανατρέξουμε και στους ορισμούς τους οποίους ε, είχαμε συμφωνήσει στο παρελθόν, που ορίζουν ποιες είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ε, και πώς διαφοροποιούνται από πλευράς ε, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, αλλά να μην τις διαφοροποιούμε μεταξύ των. Και επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς, κυρίως για όσους δραστηριοποιούνται εντός των κρατών μελών, αλλά χρειάζεται και ένα σαφής ορισμός πρέπει να διασφαλίσουμε χρηματοδότηση και θα πρέπει να το ε, συνδέσουμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τους κανονισμούς για τα αντίστοιχα ταμεία και για να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση για τον τομέα αυτό. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή χρηματοδότηση, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τη χρηματοδότηση στους κανονισμούς των ε, υφιστάμενων ταμείων. Όσον αφορά τώρα το νομικό καθεστώς, αυτή η πρωτοβουλία να υπάρχουν επισημάνσεις και να υπάρχουν καινοποιημένα κριτήρια για να μπορέσουμε να δούμε και πώς μπορούν να ε, δραστηριοποιούνται και διεθνώς αυτές οι επιχειρήσεις και φυσικά ε, και τα κριτήρια ποιοτικών υπηρεσιών ε, στον τομέα αυτό. Καταρχάς όμως θα χρειαστούμε δεδομένα επακριβή δεδομένα που να μας δείχνουν πόσο συνεισφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις στην κοινωνική ένταξη, στις κοινωνικές υπηρεσίες, ε, και θα πρέπει να αναγνωρίζει και να προβάλλεται καταλήλω αυτό ο τομέα, ο οποίο είναι πάρα πολύ απαραίτητο σε πολλές χώρες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε καλύτερο το κείμενο αυτό, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο για το κλάδο και τις διαμεθοριακές πτυχές ε, του συγκεκριμένου τομέα. Σα ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάνει άλλο το λόγο. Η κυρία Χίρς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, διότι πιστεύω με την έκθεσή του έχουμε μια πολύ καλή βάση, επί της οποίας μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχει ήδη αναφερθεί το θέμα των ορισμών. Νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια στον τομέα των ορισμών, να μην έχουμε ένα κλειστό σύστημα, να έχουμε ευελιξία, αλλά νομίζω όταν έχουμε ένα σύστημα το οποίο δίνει κοινωνικές υπηρεσίες, όπως παραδείγματος χάρη η φροντίδα των, σε παιδικούς σταθμούς, η περίθαλψη κτλ. Και έχουμε εδώ πέρα φυσικά και τους δημόσιους φορείς και τους ε, ιδιωτικούς φορείς. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τομέας, ο οποίος είναι οι επιχειρήσεις που δίνουν κοινωνική προστιθέμενη αξία, παραδείγματο χάρη δίνουν δουλειά σε ανθρώπους με αναπηρίες. Είναι σημαντικό να σταθούμε και σε αυτό το θέμα, από την ε, οπτική γωνία του επιχειρηματία ο οποίος προσφέρει έργο με αυτόν τον τρόπο. Παραδείγματος χάρη εγώ θυμάμαι ένα, ε, ένα συνεργείο για ποδήλατα στο Μόναχο το οποίο απασχολούσε άτομα με αναπηρίες και παρόλα αυτά δουλεύει πολύ καλά. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα της διαμεθοριακής πηγής και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να, να το εξάρουμε ιδιαίτερα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να μπορούν οι επιχειρήσεις να εργάζονται και σε γειτονικά κράτη-μέλη και με τον εισηγητή έχουμε συζητήσει ήδη το θέμα αυτό, αλλά ίσως θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή την ε, προσθέμενη αξία που προέρχεται και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτές οι κοινωνικού χαρακτήρα επιχειρήσεις να έχουν μια ειδική χρηματοδότηση. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα σημεία τα οποία μπορούν να καλυφθούν με τροπολογίες. Και έχουμε βέβαια μια χωριστή έκθεση για την εταιρική κοινωνική ε, ευθύνη και υπευθυνότητα, αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει ίσως να αναφερθεί στην έκθεση αυτή. Στο σημείο 16 της έκθεσης αναφέρεται αυτό ότι η κοινωνική επιχείρηση πρέπει να έχει και το χαρακτήρα της επιχειρήσεως η οποία προσφέρει ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Και αυτό φυσικά μπορεί να είναι ένα στοιχείο της γενικότερης συζήτησης που κάνουμε για τη μορφή που πρέπει να έχει μια καπιταλιστική οικονομία, να έχουμε υπόψη μας και το ποιος δουλεύει σε αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τι ακριβώς παράγουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο του ορισμού τους πιστεύω. Δεν βλέπω να θέλει κανεί. Κύριε μακκιντάερ Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τις διαβουλεύσεις με τις άλλες ομάδες. Εν γέννη υποστηρίζω τις προτάσεις της εισηγήτριας. Εν γέννη υποστηρίζουμε τις ε, καλές πρακτικές. Ε, ένα-δύο πράγματα τα οποία ίσως ε, τα είπε ήδη στον εισηγητή. Ορισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητα και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, στα αγγλικά δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των ε, δύο. Ελπίζω ότι δεν θα μπλέξουμε με τους ορισμού αυτών των δύο πραγμάτων. Επίσης, υποστηρίζω το σημείο 5, ότι οι κοινωνικέ επιχειρήσεις δεν προσανατολίζονται αναγκαστικά στο κέρδο. Και όμω στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων που παρέχουν θέσει εργασία, ε, αναπήρου, οι οποίε κατά τα άλλα λειτουργούν με εμπορικά κριτήρια. Υπάρχουν επίση επιχειρήσεις ή οργανισμοί που έχουν διεθνή χαρακτήρα. Έχουμε δίκτυα ε, τα οποία οργανώνουν πρακτικές ασκήσεις, εργαστήρια σε διάφορες χώρες. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλό θα ήταν να μην σταματήσουμε, να μην δημιουργήσουμε εμπόδια για τέτοιου είδους καλές προσπάθειες. Γιατί καμιά φορά πάμε για καλό και τελικά δημιουργούμε προβλήματα. Και μία ερώτηση στο 6. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις βεβαίως δραστηριοποιούνται σε διάφορους διαφορετικούς τομείς. Οπότε δεν κατάλαβα εδώ που κολλάει ο μη ρυθμιζόμενος ανταγωνισμός. Τι σημαίνει αυτό. Και στο 13 μου προξένεται σε εντύπωση το εξή για το ιδρυτικό, καρστερικό κλπ. Και το θέμα της ε, φορολογικής ε, αρμοδιότητας. Πέραν αυτών πάντως σύμφωνα με το κείμενο και το υποστηρίζω. Πρόεδρος, κανείς άλλος όχι. Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή, έχω και εγώ δυο τρεις παρατηρήσεις. Όσον αφορά τον τίτλο καταρχήν δεν έχουμε καταλήξει, διότι λέμε ένα σωρό διαφορετικά πράγματα εδώ, όλα κοινωνικά είναι η κοινωνική οικονομία, η ελεγγύη κλπ. Θυμίζω παλαιότερες εργασίες μας, την έκθεση το για να θυμάστε, που πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη μας. Τώρα ο χρόνος βεβαίως πιέζει, αλλά πρέπει να εκφέρουμε γνώμη επί αυτής της γνωματορής πρωτοβουλίας. Φυσικά ο εισηγητής είναι αρκετά φιλόδοξος και έχουμε και την κυρία Κόνη και την έκθεση στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Ε, μια έκθεση η οποία ανταποκρίνεται, απαντά αν θέλετε στην πρόταση του Επιτρόπου Μπαρνιέ για την δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης ειδικά για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τώρα, στην έκθεση της κυρίας βλέπουμε καλυπτόμενα στοιχεία. Και σε αυτήν την έκθεση τώρα πάλι εδώ, πρωτοβουλίας, Αντίστοιχα, φυσικά είναι καλό να στείλουμε το μήνυμα με την προϋπόθεση να μην ξανανακαλύπτουμε τον τροχό. Να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, που πηγαίνουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Αν είναι απλώς να θυμίσουμε τι κατά τα άλλα συζητούμε, η εκθέση πρωτοβουλία είναι σπάνιες και, και ακριβές θα έλεγα. Οπότε ας τις ε, χρησιμοποιήσουμε με φιδό. Εξαρτάται λοιπόν από το αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε γιατί αυτή η έκθεση. Τι θέλουμε να πούμε με μια έκθεση πρωτοβουλίας. Όμως ο εισηγητής εν προκειμένου δεν έχει, δεν έφερε σε πέρα στην ευθύνη, το ρόλο αυτών μέσα σε αυτό ακριβώς το πνεύμα. Του δίνω το λόγο αμέσως. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία, και εγώ θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσες οι προθεσμίες για τις διάφορες εκθέσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί υπάρχει και μία μορφή αλληλένδετου μεταξύ των εκθέσεων αυτών και μας δίνουν και τη δυνατότητα να δούμε την ε, διαδοχικότητα αυτών των εκθέσεων. Φυσικά όμως εγώ σε αυτή την έκθεση θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω το γεγονός ότι υπάρχουν φυσικά διαφορετικές απόψεις και εφόσον μιλάμε για κάτι καινούριο, ε, μιλάμε για ένα ταμείο επένδυσης σε κοινωνικό επιχειρήν όσο και οξύμορο να φαίνεται αυτό, Φτάνουμε λοιπόν από αυτό το τομέα μέχρι τα θέματα της κοινωνικής εταιρικής αρμοδι... Ε, Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την έκθεση εγώ θα ήθελα να ενισχύσω και όχι να αποδυναμώσω τις προσπάθειες της Κομισιόν. Ελπίζω ότι αυτό θα καταστεί δυνατό να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να τις ενισχύσουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πρώτο να προστατεύσουμε τις δομές οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί και εντηρήσουμε την πολυμορφία αυτών των φορέων που ξεκινάνε από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι συνεταιριστικά συνεργεία όπως αναφέρθηκε να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα διατηρηθεί η πολυπικιλία αυτών και δεύτερον να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για τέτοιες επιχειρήσεις σε κοινωνικό επίπεδο και ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι σημαντικό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν ή αν θέλετε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό που υπάρχει και να το κάνουμε χρησιμοποιήσιμο. Επομένως να βρούμε την κατάλληλη κανονιστική ρύθμιση η οποία αντί να περιορίσει θα επιτρέψει την ελεύθερη άνθηση και αναδίπλωση όλων αυτών των δυνατοτήτων κοινωνικού επιχειρήν που θα πρέπει να προστατευτούν και να ευνοηθεί η ανάπτυξή τους. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μια κοινή κατανόηση για αυτό το θέμα και ελπίζω θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Οπότε η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 5 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. 20 Ιουνίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Οι συμβιβαστικές θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν στις 10 Ιουλίου. Πάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 23, έκθεση της κυρίας Μακιντήρ ή Μακιντάιρ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα καθώς και τις προοπτικές στον εμπορικό τομέα πρόκειται για τα σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο προορίστηκε για την Επιτροπή Ήτρε. Σας δίνω το λόγο κύριε Μακιντάιρ. Thank you very much, Madam Chairman. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όπως εξηγήσατε μόλις, αυτή είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης για την ε, έκθεση της Επιτροπής ε, Ήτρε, που είναι μια ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ανταγωνιστικότητα και τις εμπορικές τους προοπτικές ως Επιτροπή Απασχόλησης προφανώς επικεντρωνόμαστε στην πλευρά της απασχόλησης. Να ευχαριστήσω πολύ τους κοιόδες συντάκτες, διότι ε, μου έδωσαν πολύ καλές προτάσεις στις αρχικές μου εισηγήσεις και θα ήθελα να τις συμπεριλάβω και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαζόμαστε υπ' αυτό το πνεύμα. Όπως γνωρίζουν όλοι, επειδή ούτως ή άλλως ε, το μέγιστο μιας γνωμοδότησης είναι 1500 χαρακτήρες, δεν μπορούμε να περιλαμβάνουμε όλα όσα θα επιθυμούσαμε. Προσπάθησα λοιπόν να είμαι λακωνική και να χρησιμοποιήσω αυτή τη γνωμοδότηση για να δημιουργήσω τα θεμέλια από τα οποία θα οικοδομήσουμε όλοι μια ακριβή και συνεκτική γνωμοδότηση ήλπιζα να μπορέσω να συμπεριλάβω και την ιδέα της κυρίας Ρέντερ για το One Stop Shop, αυτή την ενιαία θηρίδα. Δεν νομίζω ότι με ακούει. Ελπίζω λοιπόν να μου καταθέσει και σχετική τροπολογία για να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν θα σας απασχολήσω με αυτά εδώ, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Αλλά το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχουν 90 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Το 30% προέρχεται από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και νομίζω ότι αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Συνεργάστηκα με τον εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή και προσπάθησα να μην επαναλάβω τα όσα λέει αυτό, αλλά να είναι μια συμπλήρωση γνωμοδότηση και ελπίζω να υποστηρίξει και το σημείο 9 τη γνωμοδότησής μου. Δηλαδή, να διευκολύνουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, σε ένα ενισχυμένο κείμενο, ε, σε ένα ενισχυμένο πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. δεν θα λέμε ότι εξαιρούνται, αλλά θα λέμε ότι κάθε φορά θα πρέπει να χρησιμοποιείται η νομοθεσία για αυτές τις μικρές επιχειρήσεις και ιδίω τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Θα ήθελα να σχολιάσουν και οι σκιώδεις εισηγητές και προσβλέπω στην ε, συνεργασία μαζί τους και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Τίερ, συνάδελφοι. Η Εύελιν Ρίκνερ, η εκπρόσωπος των σοσιαλιστών, δυστυχώς απουσιάζει και μου ζήτησε να παρουσιάσω εδώ τη δική της γνωμοδότηση. Λέει τα εξής κυρία Ρέγνερ. Θέλω κυρίως καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί όλοι οι ισχυώδεις εισηγητές παρέστησαν σε μία συνάντηση. <clears throat> Έχει κάθε εμπιστοσύνη ότι θα, υπάρξει, θα υπάρξουν περαιτέρω επικοδομητικές συναντήσεις και θα καταλήξουμε σε μία, σε μία καλή απόλυξη. Για την γνωμοδότηση, ο στόχος μας είναι, ανεξάρτητα από πολιτικές παρατάξεις, να δημιουργήσουμε ένα έφορο πλαίσιο εργασίας και οι προτάσεις της κυρίας Ιντάερ θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτόν τον σημαντικό εργοδότη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει ε, πρόοδος και επιτυχία και των εργοδοτών και της οικονομίας γενικά. Φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται από την ικανοποίηση των εργαζομένων και το πρόσφορο χαρακτήρα του, του εργασιακού ε, πλαισίου από την πλευρά των σοσιαδημοκρατών το να υπάρχει μονάχα προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημαίνει ότι δεν δίδουμε τη δυνατότητα στους εργαζομένους να παίξουν το ρόλο τον οποίο πρέπει να διαδραματίσουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Αναφέρεται πάρα πολλές φορές ότι το... η διατήρηση των κανόνων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει ότι θα οδηγήσει σε προβλήματα για τους εργαζομένους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να μην εξαιρεθούν από τις προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Θέλω να τονίσω ότι αυτές οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελάχιστες προδιαγραφές. Επομένως δεν μπορούμε ποτέ, ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας επιχείρησης, να τους δώσουμε εξαιρέσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε τους εργαζόμενους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να <clears throat> εκτίθενται σε μεγαλύτερους κινδύνους από αυτούς των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό είναι μια πολύ βασική αρχή που ελπίζει ότι θα μπορέσει να βρει τη συμφωνία του μεγαλύτερου μέρους της Επιτροπής μας. Σε πολλές χώρες, όπως η Αυστρία, είναι οι 90% των επιχειρήσεων μικροεπιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μέχρι 10, μέχρι 10 εργαζομένους. Δεν θα πρέπει να έχουν εξαίρεση και να μην μπορούν να μην υποχρεωμένους να τηρούν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και την προστασία της υγείας τους. Η γνωμοδότηση της κυρίας Μακριντάε δεν λαμβάνει επίσης απόλυτα την ε, μεγάλη σημασία σε κοινωνικό επίπεδο των θετικών προτύπων εργασίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Εμείς ως, επιχει... ως ε, Επιτροπή Απασχόληση θα πρέπει να θέσουμε στο εστιακό σημείο το πλαίσιο εργασίας και την προστασία των εργαζομένων και να εξασφαλίσουμε την μεγαλύτερη δυνατή προστασία των εργαζομένων και να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Μπενιό και μετά ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή. Δηλαδή τα πήγαμε εξαιρετικά μέχρι και σήμερα. Πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι απαραίτητε για να πάμε μπροστά, να αντιμετωπίσουμε την τελμάτωση της οικονομίας. Φυσικά θα προκύψουν κάποιες πολιτικές διαφορές ε, προκειμένου, αλλά εν γέννη προκύπτει συμφωνία ότι πρέπει να βελτιώσουμε βέβαια το περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον για μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει να απλουστεύσουμε μεταξύ άλλων το λεγόμενο διοικητικό φόρτο, χωρίς να μοιέσουμε την κοινωνική προστασία των εργαζομένων. Μπορούν να γίνουν και τα δύο με προσοχή. Μπορούμε λοιπόν να απλουστεύσουμε, όπως είπα, τις διαδικασίες, διατηρώντας υψηλά επίπεδα τους κανόνες απασχόλησης. Η ασφαλή και η υγεία. Ας πούμε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Το αντιμετωπίσαμε με αυτόν τον τρόπο και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Διευκολύναμε δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να υπονομεύσουμε τα θέματα, τους κανόνες ασφαλεία και υγείας. Εγώ προέρχομαι από μια πολύ μικρή επιχείρηση, ξέρω το χώρο και ξέρω τι σημαίνει ένας άνθρωπος να είναι υπεύθυνο για τα πάντα. Δεν είναι όπως σε μια μεγάλη επιχείρηση που έχετε ολόκληρα τμήματα και διευθύνσεις για να ασχολούνται με, το, με τον κάθε νόμο. Όχι, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις ένας άνθρωπος κάνει τα πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Συμφωνώ όμω κατά άλλα ότι δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τους κανόνες ασφαλείας και υγείας. Γνωρίζω τους περιορισμούς αυτής της γνωμοδότησης, γιατί είναι της ΙΤΡΕ κυρίως ε, βεβαίως αρμοδιότητα και ξέρω και το όριο σε λέξεις που αντιμετώπισε η κυρία Μακεντάιρ. Έχουμε τροπολογίες, συνεπώς, για να αξιοποιήσουμε τις ήδη καλές προτάσεις και να βελτιώσουν και το περιεχόμενο. Δεν θέλω να υπερβώ τα όρια της εντολής μας, αλλά η πρόσβαση σε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για παράδειγμα, είναι σημαντική. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι κινήσεις που θα διευκολύνουν τις μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει να μεγαλώσουν, να προσλάβουν προσωπικό κλπ. Αυτά προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία και με τι άλλε ομάδε για να στηρίξουμε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο ευχαριστώ. Άλλο κανεί που θέλει το λόγο. Ο κύριο Μπέκερ καταρχήν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία όπως είναι φανερό έχει ένα πάρα πολύ συνεργατικό και επικοδομητικό τρόπο εργασίας. Για το ίδιο το περιεχόμενο της έκθεσής της, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια αριθμητικά στοιχεία τα οποία έχουν μια επιτακτική λογική. Ξέρουμε ότι είναι 23 ε, επιχειρήσεις στην Ευρώπη, δηλαδή το 90% όλων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η σημασία αυτών των επιχειρήσεων στο ευρωπαϊκό οικονομικό στερέωμα, ιδίω όταν γνωρίζουμε ότι ακριβώς είναι ο τομέας ο οποίος είναι ο πιο ανθεκτικός στην κρίση, πολύ περισσότερο από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν σαφές όπου ότι μπορούμε και πρέπει να ευνοήσουμε τις ε, συνθήκες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως ελέγχθη αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της προστασίας και της ε, <clears throat> υγείας των εργαζομένων, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια ελάφρυνση του κανονιστικού πλαισίου και της γραφειοκρατίας, γιατί όπως ξέρουμε αν η κάθε μια από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις προσλάβει ένα εργαζόμενο, θα έχουμε 23, 23 ε, εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Εντάξει, αυτό είναι λιγάκι μαύρο-άσπρο, είναι κάπως ε, σχηματικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην απασχόληση και στην οικονομία. Για μένα <clears throat> το θέμα του, της μικροχρηματοδότησης, έχουμε ήδη το παράδειγμα του Εράσμου για τους νέους, του Εράσμους για τους νέους εργαζόμενους, και επιχειρηματίες και είναι σημαντικό να προωθήσουμε αυτή την διτή μορφή κατάρτισης δίνοντας τις κατάλληλες ευκαιρίες και πληροφορίες και ελπίζω θα έχουμε και πολύ καλή συνεργασία με την συγγετρία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σωστό ότι ήδη με την εισηγήτρια έχουμε πολλά κοινά σημεία σε επίπεδο περιεχομένου. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν αντανακλώνται πλήρως στο κείμενο από αυτά τα οποία αναφέραμε. Νομίζω ότι έγινε σαφές και από αυτά που διάβασε η κυρία Στάινρουκ από το κείμενο της κυρίας Ρέγνερ. Νομίζω ότι ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Δεν είμαστε η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, η Επιτροπή Ήτρε, η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει τα θέματα γενικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα ποια είναι η πτυχή της ε, απασχόλησης και οι κοινωνικές πτυχές που συνάπτονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο θα καταθέσουμε ορισμένε τροπολογίες και κυρίως για τα θέματα τα οποία είναι της αρμοδιότητας της δικής μας Επιτροπής. Θα ήθελα να σας το πω αυτό εκ των ε, προτέρων και αυτό είναι φανερό και από την ε, γραπτή δήλωση της κυρίας Ρέγνερ Προβλέπουμε βέβαια ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο κείμενο, αλλά τονίζουμε ότι τα θέματα αυτά που μας ενδιαφέρουν προ το παρόν ελείπουν από το κείμενο. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω πια κάποιον ο οποίο να ζητάει το λόγο. Θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Μακιντήρ. Να ευχαριστήσω όλους τους και οδησχύτες για τα σχόλιά τους. Κύριε Στάνερ, παρακαλώ να μεταφέρετε στην κυρία Ρέγνερ ε, κάποια από τα σχόλια που θα ακούσετε εδώ. Γιατί, ε, κοιτάξτε, εμεί ε, παλεύουμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων σε οποιοδήποτε τομέα. Γι' αυτό και στο σημείο 8, αφού μιλήσαμε με την κυρία Βέγνερ, γράψαμε εδώ για την ασφάλεια, την υγεία και την ισότητα. Εδώ προσπαθούμε ακριβώς όχι να υπονομεύσουμε όλα αυτά, αλλά να κάνουμε πιο εύκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με την νομοθεσία. Όχι το αντίθετο. Ούτε προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διαφοροποίηση μεταξύ εργαζομένων στη μία κατηγορία σε σχέση με μια άλλη. Απλώ για έναν άνθρωπο μόνο του είναι πολύ πιο δύσκολο να συμμορφώνεται με την νομοθεσία έτσι όπω έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό, αυτό που είπε η κυρία Σρέντερ για το One Stop Shop, το κέντρο εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να το βάλουμε και το αναφέρω εδώ, όπως είδατε. Αλλά λόγω του ορίου των λέξεων ε, περιορίστηκα και δεν το είδατε στο κείμενο. Άκουσα όλα τα σχόλια και περιμένω ανυπομονησία της τροπολογίας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε μια έκθεση, σε μια γνωμοδότηση μάλλον, με την οποία θα μπορέσει να συμφωνήσει όλη η Επιτροπή. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Οπότε, προθεσμία αρχή ξεκινάει 5 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Θα τη συζητήσουμε στις 20 Ιουνίου. Ψηφίσουμε την επόμενη και η Ήτρε θα ψηφίσει στις 11 Ιουλίου. Κατά επέκταση αυτή τη συζητήσεω, υποβάλλω σχέδιο προφορική ερώτηση με έτοιμα προφορικής απάντησης και σχέδιο σχεδίου πρότασης ψηφίσματος, το οποίο συνοδεύει την ερώτηση αυτή. Πρωτοβουλία των συντονιστών όσον αφορά τις επιπτώσεις επί της απασχόλησης λόγω, χάρη στην μείωση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ. Η κυρία Μακεντάιρ δούλεψε στη σκιά της Ήτρε βεβαίω, λαμβάνοντας υπόψη κείμενα επίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα οποία φύγεται η κοινωνική διάσταση, ε, αλλά όχι όμως επαρκώς. Βάσει αιτήματος των έχω την ευθύνη να σας παρουσιάσω το σχέδιο ερώτησης και το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος. Ως προς την ερώτηση, την προφορική ερώτηση που θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια κοινή ε, συζήτησης με την Επιτροπή Ήτρε για τις μικρομεσαίες θα επιμείνουμε στο ερώτημα περί του κατά πόσον η μείωση του κανονιστικού φόρτου που θα είναι υπέρ των ΜΜΕ θα έχει ως αποτέλεσμα την επιδίνωση των επιπέδων κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων που εργάζονται για ΜΜΕ. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο είναι το εξής. Πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να σωματώσουν με βέλτιστο τρόπο μισθωτούς στο οργανόγραμμά του και να εκπροσωπούνται παρκώς. Με αφορμή αυτό το ερώτημα, ρωτάμε την Κομισιόν σε ποιο βαθμό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση. είναι ερώτημα που είχαμε απευθύνει στην αρχή της εντολής. Στο σχέδιο ψηφίσματος προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα ζητήματα που θίξαμε. Καταρχήν για να υπενθυμίσουμε το πρόβλημα των μικρομεσαίων, την ανάγκη ευελιξία στην απασχόληση. Εκφράζουμε την λύπη μας διότι πολύ λίγα κράτη-μέλη λαμβάνουν υπόψη τους τις μικρομεσαίες όταν νομοθετούν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που είχαμε πει είναι πριν από την έγκριση ή οδήποτε νόμου να μελετάτε οι επιπτώσεις που έχει νέα νομοθεσία στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο θα είχε ενδεχομένω ως αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να αποκλείονται όταν αυτό δεν απαιτείται από την εφαρμογή του ενός του νόμου. Δηλώνουμε επίσης την υποστήριξή μας στα δικαιώματα των εργαζομένων και σε υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασία. Επίσης, υποστηρίζουμε την υλοποίηση των ε, συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Κατόπιν πρωτοβουλίας της ε, Επιτροπής μας ζητούμε να δημοσιευτούν οι 10 πιο γραφειοκρατικές αποφάσεις για τις ΜΜΕ. Καλούμε την Κομισιόν επίσης να δημιουργήσει ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης για τις μικρομεσαίες και να δημιουργήσει και ένα φόρουμ καλών πρακτικών. Ως προς το θέμα της εκπροσώπησης και δι των ανεξαρτήτων εργαζομένων είναι κάτι που πρέπει επίσης να φροντίσουμε στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρωτοβουλία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκολύνει τη χρηματοδότηση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, πολύ ενδιαφέρον για τι μικρομεσαίες. Και τέλος, δηλώνουμε ότι θεωρούμε ότι εν γέννη στα κράτη-μέλη το θέμα της επιχειρηματικότητας και των σχετικών γνώσεων πρέπει να προωθηθεί και μέσω της παιδείας, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες υπέρ της εκμάθησης ξένων γλωσσών για τους υπαλλήλου μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Πολύ σημαντικό για την, την κλίμακα. Προτείνουμε επίση οι διατάξει της μικρομεσαίας να ισχύουν και του ανεξαρτήτους εργαζομένους. Είναι ένα θέμα το οποίο το παντούμε και στη συζήτηση περί του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και Σάρκιν. Και βεβαίως τέλος υπενθυμίζουμε το ζήτημα του άρθρου 9. Βλέπετε λοιπόν με περισσότερες λεπτομέρειες την κεντρική ιδέα που διατρέχει το ψήφισμα. Ο στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υπονομεύσουμε την νομοθεσία που προστατεύει τους εργαζόμενους και την δυνατότητα διαπραγμάτευσης που έχουν στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου. Αυτά ήθελα να σας παρουσιάσω. Ο κ. Κλάρκ τώρα ζήτησε τον λόγο και μέσω ο κ. Πενιό. Ο κ. Κλάρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ και με την έκθεση και με την πρόταση προφορική ερώτηση και τι χαιρετίζω και τι δύο. Έχετε δίκιο κύρια Πρόεδρε. Η παιδεία διδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πτυχή αυτή. Αλλά νομίζω ότι το όλο θέμα της συνδρομής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ξεκινά από τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτό θα πρέπει να προτείνουμε και θα πρέπει ε, να είναι αυτό, διότι είναι το μεγαλύτερο πρόσκομα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις πιο μικρές, ε, δεν μπορούν να προχωρήσουν τις δουλειές τους, δεν μπορούν να ασκήσουν το έργο τους και φυσικά αναγκάζονται να απολύσουν εργαζομένους η έκθεση ζητά από τις μικρές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ε, ε, ανεξάρτητες ε, ομάδες εκπροσώπων κλπ. κλπ. Σε κάποιο βαθμό αυτό θα ε, είναι χάσιμο χρόνο για τους μικρούς επιχειρηματίες, διότι θα πρέπει να σπαταλούν το χρόνο τους, να συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες των εκπροσώπων, ενώ θα, στην πραγματικότητα θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει, ίσα ίσα θα τους προσθέσει επιπλέον άχθος και νομίζω ότι αυτό θα είναι εις βάρος τους τελικά. Προχωρώντας όμως, δύο φορές και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια έχω ρωτήσει τον Επίτροπο Άντορ τι σκόπευε να κάνει προκειμένου να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μειώσουν τη γραφειοκρατία και, τις, και το κανονιστικό φόρτο. Και ποτέ δεν μου απάντησε κάτι σαφέ. Πολλό δε μάλλον που τώρα ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόσο, είπε πριν από δύο χρόνια ότι η γραφειοκρατία ε, ουσιαστικά στραγγαλίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξακολουθεί να το κάνει. Να σας παραπέμψω λοιπόν κυρία Πρόεδρε στο, τμήμα, στο σημείο 3 της προφορικής σας ερώτηση που λέτε ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή προκειμένου να παρακολουθήσει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην κοινωτική χρηματοδότηση και να αναφέρει τα σχετικά αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο. Να το επεκτείνουμε λίγο αυτό, ατύπως, ουσιαστικά ρωτάμε αν θέλει σοβαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δι τις πολύ μικρές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα μπορέσετε κάλλιστα να συνεισφέρετε όταν θα ε, προσπαθήσουμε να περάσουμε αυτή την πρόταση μέσω τροπολογιών. Ο κύριος Νιόν, σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας περιλαμβάνει αρκετές καλές ιδέες και συμφωνώ. Έχει και πολλά στοιχεία που τη συνδέω με τις προηγούμενες εκθέσεις. Λίγο πολύ στα ίδια θέματα αναφερόμαστε. Με απογοήτευσε λίγο η απάντηση του Επιτρόπου Άντορ την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι είχε αμυντική στάση, ιδίως για τα κανονιστικά ζητήματα αλλά όπως είπα νομίζω ότι σε αυτή την έκθεση ε, βλέπουμε κάποια θετικά στοιχεία και νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε θετικές ιδέες, ε, ε, κατόπιν συζήτησης, μπορεί να μην συμφωνούμε ίσως όλοι, αλλά νομίζω ότι προκύπτουν αρκετές καλές ιδέες από αυτό το κείμενο. Κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε ίσως είναι και ε, το πώς νιώθει το κάθε κράτο μέλος για το ε, κανονιστικό φόρτο. Ξέρω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ιδίω ο τύπος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος ε, μπορεί να πάρει μια κανονιστική ιδέα και αρχίζουν από εκεί και πέρα να τις χρησιμοποιούν παντού. Ε, μπαλάκι. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν τι γίνεται με το κανονιστικό πλαίσιο και να λάβουμε υπόψη ότι είναι και διαφορετικές οι συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος. για την κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους, όπως έχω πει και στο παρελθόν, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη ζωφερή εικόνα ότι η απλούστευση της νομοθεσίας είναι αυτομάτως και επιδείνωση της κατάστασης των εργαζομένων. Εάν γίνουν όλα αυτά προσεκτικά, δεν χρειάζεται αυτόματα να οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, ίσως θα έπρεπε να βελτιώσουμε τη συνεισφορά των μικρών επιχειρήσεων, δηλαδή πώς μπορούν να συνεισφέρουν στους κοινωνικούς εταίρους όχι μόνο τους αγνοούμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πολύ συχνά τους αγνοούν και τα ίδια τα κράτη-μέλη ε, στις διαδικασίες διαβούλευσης. Όταν γίνονται διαβουλεύσεις, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των συνδικάτων και φυσικά και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, αλλά πολύ συχνά οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν λόγο. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους τομείς που συνεισφέρει ε, πολύ στην ε, δημιουργία νομοθεσίας, ε, την οποία μπορούν πολύ εύκολα να εφαρμόσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά όχι τόσο εύκολα οι μικρές. Το να περιλάβουμε λοιπόν και αυτές τις μικρές επιχειρήσεις εντός του πλαισίου είναι εξαιρετική κατά την άποψή μου και θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Για την παρατήρηση τώρα του κυρίου Κλάρκ για τη δημιουργία φορο... αντιπροσωπευτικών φορέων. Νομίζω ότι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν ομάδες εκπροσώπων ε, μικρών επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους ε, που δικαίως έχουν δημιουργήσει ομάδες εκπροσώπων. Υπάρχουν πολλά συνδικάτα τα οποία ακούμε τακτικώς όταν προτείνεται κάποια νομοθεσία που τους αφορά. Δεν είμαι βέβαιος τι προσθέτει αυτό. Μήπως ε, σε κάποια κράτη-μέλη ε, ήδη συμβαίνει αυτό που προτείνουμε. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσει, ε, τι ακριβώς εννοείται με αυτούς τους ε, αντιπροσωπευτικούς φορείς. Θα προσπαθήσω να καταθέσω και σχετικές τροπολογίες και προς την, ε, για την προφορική ερώτηση και για το ψήφισμα και ελπίζω να θεωρηθούν αποκοδομητικές και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε περαιτέρω για το θέμα αυτό και να έχουμε ένα καλό έγγραφο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία, και κυρία Μακιντήρα. Αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό για μένα σε αυτό το θέμα να εξετάσουμε και το έγγραφο της Κομισιόν που δημιουργήθηκε από τη βάση της εκθέσεως Στόιμπερ για τα θέματα της ε, αφιοκρατίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ε, ποιότητα της εργασίας και τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα οποία για μένα έχουν πολύ μεγάλη αξία από τη λεγόμενη ελάφρυνση από τη γραφειοκρατία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η οδηγία για την ε, απόσπαση των επιχειρήσεων ε, θα πρέπει, η ιδέα ότι θα πρέπει να μην ισχύει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά στους τομείς που υπάρχουν μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημαίνει αυτό ότι δεν θα υπάρχει καμία απολύτως προστασία για τους εργαζόμενους στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει αυτή η προστασία. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να υποστηρίξω μια τέτοια λύση γιατί αυτή θα σήμαινε ότι θα είχαμε ένα μαζικό κοινωνικό dumping και τα 95% των επιχειρήσεων θα έχουν πια απόλυτη απώλεια προστασίες και θα γίνει πραγματικότητα το dumping. Θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να κάνουν ε, dumping αυτές οι επιχειρήσεις χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά θα συμβάλλουν αυτές οι επιχειρήσεις στην, αθέμητη, σε αθέμητο ανταγωνισμό σε σχέση με τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε μια περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν την νομοθεσία, αλλά οι, αυτές που έρχονται από απ' έξω δεν θα είναι υποχρεωμένες να κάνουν κάτι τέτοιο. Πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό πολύ προσεκτικά σε σχέση με το θέμα αυτό και πρέπει αυτή η προβληματική να βρεθεί στο κέντρο της προφορικής ερώτησης και του ψηφίσματος. Σας ευχαριστώ, λέει Κυρία Μακιντία. Και εγώ, όπως και άλλοι, εκφράζω την ικανοποίησή μου για αυτό το σχέδιο πρόταση ψηφίσματος. Και ζηλεύω γιατί καταφέρατε να στριμώξετε εδώ περισσότερα πράγματα από ό,τι σε μια γνωμοδότηση. Σίγουρα θα προκύψουν τροπολογίες, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ε, πνεύμα επικοδομητικό. Βεβαίως. Μ' αρέσει αυτό που λέτε εδώ, ότι περισσότερες ε, μικρομεσαίες σημαίνει επιχειρηματικότητα, διότι η αυτοπασχόληση Μεταξύ άλλων συμβάλλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην Ευρώπη. Κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στις ε, μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και την ανάγκη να δημιουργήσουν όργανα εκπροσώπησης. Ο οποίος ε, είναι στον τομέα. Εγώ ας πούμε ήμουν σε μια συνομοσπονδία, ομοσπονδία πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ναι, ε, υπάρχουν, υπάρχουν τέτοια πράγματα και συμφωνώ. Όμως υπάρχουν ήδη πολλά τέτοια όργανα σε διάφορες χώρες και το μόνο που δεν θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε επικαλύψεις και παραλήψεις. Λοιπόν, ναι, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών. Σύμφωνα με τα περισσότερα εδώ, εξαιρετικά σχόλια, εξαιρετική δουλειά. Προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία επί Ευχαριστώ. Ο κ. Πρόεδρε. Μήπως εδώ συζητούμε κάποια ουτοπική πραγματικότητα, μήπως ονειρευόμαστε. Μιλάμε για κοινωνικό διάλογο στις μικρομεσαίες. Στις μικρομεσαίες δεν υπάρχει συνδικάτο. Ε, δεν χρειάζεται μάλιστα. Θα λέει κανείς, γιατί εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπω κάθε μέρα. Μετά λέτε δημιουργία θέσεων εργασίας. Μα η αγορά δημιουργεί τις θέσεις εργασίας. Όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις απολύουν, όταν μεταγκαθίστανται εκτός Ευρώπης, ποιος θα αγοράσει τις υπηρεσίες τους. Μπορώ να αγοράσω οτιδήποτε μόνο όταν έχω έσοδα, μόνο όταν έχω ένα μισθό. Αυτό μου φαίνεται τώρα όνειρο θερινής νυχτός. Για ποιου μιλάτε, τι, θέλετε να κάνουν, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι αυτά πατώμεθα. Φέρτε εδώ τους επιτρόπους, Σπίτλα κάθε φορά που προσπαθούν να κάνουν κάτι, τα κράτη-μέλη αρχίζουν να ουρλιάζουν περί επικουρικότητας κλπ. Αυτό το οποίο θέλουν είναι νομοθεσία που δεν θα εφαρμόζεται, νομοθεσία που δεν θα λειτουργεί και θα επιτρέπει τα πάντα. Σας ευχαριστώ για αυτές τις παρατηρήσεις. Βέβαια υπάρχει αυτό, αυτή η διτή μορφή αντιμετώπισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δούμε και αυτή η πλευρά των πραγμάτων. Όταν τίθεται το θέμα της ανταγωνιστικότητας στα κράτη-μέλη μας. Και μετά κραδένουν την επικουρικότητα τα κράτη-μέλη, όπως είπε και ο τελευταίος ο μιλητής, όταν τα θέματα αυτά τους δημιουργούν προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει να μας υπενθυμίσει και να υπενθυμίσει τους άλλους ποια είναι τα θεμέλια του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Γιατί αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η βάση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, αλλά δεν λέμε τίποτα για τα κοινωνικά θέματα, τότε θα δημιουργήσουμε ε, θύλακους ανομίας για τους εργοδότες οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς κανένα περιορισμό. Και δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Το θέμα της πληροφόρησης, το θέμα του κοινωνικού διαλόγου, των συλλογικών συμβάσεων, των διαπραγματεύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τίθεται διαφορετικά από ότι για μια μεγάλη επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι οι συνδικαλιστικές δομές και οι δομές του κοινωνικού διαλόγου έχουν γεννηθεί μέσα από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά επειδή τώρα προχωρούμε προς μια άλλη μορφή επιχειρήσεων, θα πρέπει να θέσουμε αυτό το ερώτημα και να δούμε πώς μέσα σε αυτό το νέο οικονομικό πλαίσιο μπορούν να αντιμετωπίζονται τα κοινωνικά ζητήματα. Εξού και η πρόταση στην οποία εγώ επανέρχομαι και για την οποία θα έχετε φαντάζομαι τροπολογίες και για την οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Μπενιό, να υπάρξει δηλαδή η αναγνώριση ανεξαρτήτων εκπροσωπευτικών φορέων. Είναι ίσως ένας καινοτόμος τρόπος να θέσουμε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. Το καταλαβαίνω. Αν δεν θέσουμε όμως το θέμα επιτάπτως, αν δεν δώσουμε τις απόψεις μας, τίποτα δεν θα γίνει. Ανεξάρτητα λοιπόν από όλα αυτά τα θέματα, να γίνουν πραγματικότητα αυτά που λέμε για την πράσινη οικονομία, για την κοινωνική οικονομία, για την βιώσιμη οικονομία, αν θέλουμε να γίνουν πραγματικότητες όλα αυτά, δεν αρκεί να κάνουμε μεγάλους λόγους στην ε, Ρώμη, στο Παρίσι, στο Ελσίνκι και μετά τίποτα. Πρέπει να κάνουμε και επιτόπου τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι κοινωνικοί φορείς να υλοποιήσουν αυτή τη στρατηγική. Πάρτε λοιπόν το θέμα το, της κατασκευαστικής ε, βιομηχανίας, της ανακαίνησης των κτηρίων και να λέμε ότι πρέπει και να χρησιμοποιούνται περισσότερο υλικά τα οποία να έχουν αηφόρο οικολογικό, οικολογικά χαρακτήρα. Αν τώρα η εκπαίδευση των τεχνητών και των μικρών επιχειρήσεων που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα αυτό δεν είναι σωστή, τότε θα αποτύχουμε. Ανεξάρτητα λοιπόν από το θέμα το κοινωνικό, το θέμα της κατάρτισης και επομένως της ε, διάρθρωσης του ιστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να τεθεί. Πιστεύω ότι αυτά είναι ζητήματα που μπορούμε να συζητήσουμε μέσα από αυτή την έκθεση και το ψήφισμα. Και συμμερίζομαι αυτά που ελέγχθησαν για την έκθεση Στόιμπορ, η οποία ουσιαστικά, όπως είπε η κυρία Σουέντερ, ζητάει να υπάρξει μια εξαίρεση από την εργασιακή νομοθεσία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει όμως να δείξουμε πραγματικά μία εφευρετικότητα για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τις δομές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις συνθήκες εφαρμογής του κοινωνικού δικαίου και του δικαίου εργασίας. Και παράλληλα με αυτά που είπε η κυρία Μακκιντήρ στη δική της ε, έκθεση, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Κυρία λοιπόν Μακιντήρ, δεν πιστεύω ότι πρέπει να γιατί με τις τροπολογίες αυτές μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη ισορροπία. Σήμερα ο κανονισμός δεν μας δίνει όπλα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσετε να βελτιώσετε αυτή την κατάσταση. Εγώ Ανοίγω τώρα την ε, ε, προθεσμία τροπολογιών εν παραλίλω στη δική μου έκθεση και την έκθεση της κυρίας Τίερ που πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα. Στις 5 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι η εξέταση θα γίνει στις 20 Ιουνίου και η ψηφοφορία αν θέλει ο Θεός στις 21. Περνάμε τώρα σε ένα σημαντικό σημείο της ημέρησης διαταξής μας διότι πρόκειται για την έκθεση Ζίπελ για την πρόταση οδηγίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και Κοινοβουλίου για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων και αυτή βέβαια είναι στα χέρια της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και εμείς είμαστε γνωμοδοτική επιτροπή. Κυρία Ισηγήτρια, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε γνωμοδότησή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία διατύπωση την οποία <clears throat> έχει θέσει και η Κομισιόν στην, εισαγωγική, στην εισαγωγή αυτής της, ε, του νομοθετήματος ότι η διαδικασία σύναψης συμβάσεων μπορεί να υποστηρίξει κοινωνικούς στόχους και τους στόχους της ε, Ευρώπης 2020 και αυτό σημαίνει όχι μόνο περιβαλλοντικούς στόχους αλλά και στόχους κοινωνικούς. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σωστή προσέγγιση αλλά πρέπει να πω ότι η ίδια αυτή προσέγγιση δεν βλέπω να αντανακλάται πλήρως στα άρθρα της ε, πρότασης της Κομισιόν και γι' αυτό νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διατύπωση αυτού του νομοθετήματος. Ένα μεγάλο τμήμα των ε, δημοσίων προϋπολογισμών δίδεται για δημόσιες προμήθειες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πραγματικό μοχλό με τον οποίο μπορούμε να κινήσουμε τα νήματα προς την κατεύθυνση της αηφορίας της οικονομίας και αυτό θα έχει μεγάλες θετικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκομένους. Έχω αναφερθεί ιδιαίτερα στα κοινωνικά κριτήρια στη γνωμοδότησή μου και την ανάγκη να τηρηθούν οι κοινωνικοί κανόνες και οι κανόνες στο χώρο εργασίας, γιατί αυτό είναι και η αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής. Να στάθω σε ορισμένα σημεία εντάχει. Καταρχήν, το κριτήριο του χαμηλότερου κόστους θα πρέπει να διαγραφεί, γιατί αυτό σημαίνει πολλές φορές η απονομή γίνεται απλώς και μόνο με κριτήριο το κόστος. Δεν είναι αυτός ο πιο υπεύθυνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη, το καλύτερο όφελος σε σχέση με κόστος για τα χρήματα του δημοσίου τομέα. τα, τα θέματα της προστασίας και της ε, αξίας σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο πρέπει να αναφέρονται επακριβώς. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την ανάγκη να τονίζεται η σημασία του σεβασμού διεθνών ε, συμφωνιών όπως και του διεθνούς δικαίου και των συλλογικών συμβάσεων. Ιδίως όταν πρόκειται για διαμεθοριακού χαρακτήρα συμβάσεις και επίσης θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το παράτημα της Σύμβασης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτός ο οποίος προσκαλεί σε σύναψη σύμβασης θα πρέπει στις τεχνικές προδιαγραφές να σέβεται και τα, τα κοινωνικά δικαιώματα και στα κριτήρια ε, στις προδιαγραφές που αναφέρονται, αλλά και στα κριτήρια επιλογής, όπως παραγωγής χάρη, εκπαίδευση, κατάρτιση κτλ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια επιλογής δεν θα πρέπει να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, απλώς έχουν διαφορετική μορφή. Το ένα είναι απόλυτες απαιτήσει και το άλλο είναι κριτήρια επιλογής, όπως είπαμε προηγουμένως. Και επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε περίπτωση υπεργολαβίας η αλυσίδα ευθύνης μεταξύ του κύριου αναδόχου και των υπεργολαβικών φορέων ιδίω ότι πρόκειται για τις προδιαγραφές για τα κοινωνικά θέματα και το εργασιακό δίκαιο και επίσης να, ε, μέσα στα πλαίσια ενός περιορισμού των καθέτων υπεργολαβιών. Η παροχή υπηρεσιών που έχει να κάνει με άτομα θα πρέπει να προστατεύεται ιδιαίτερα, θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση εξασφάλισης της απαραίτητης ποιότητας και θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι κανόνες στον κοινωνικό χαρακτήρα και τον ε, χώρο της εργασίας, ώστε να μπορούμε με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει αυτή η απαραίτητη λειτουργία. Θέλω τέλος να τονίσω ότι είναι απαραίτητο για να υπάρξει σωστή εφαρμογή αυτής της οδηγίας να σταθούμε και στα θέματα της διακυβέρνησης. υπάρχει πάντα στη διαδικασία αυτή των, της σύναψης συμβάσεων και όταν παρατηρούνται προβλήματα θα πρέπει να υπάρχει ένα μητρό στο οποίο καταγράφονται αυτές τις δυσκολίες, το οποίο να είναι προσβάσιμο ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα συστήματα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν και η παρακολούθηση για την εφαρμογή των προδιαγραφών, ιδίω σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα εργασίας και να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μια δημόσια εποπτική αρχή η οποία θα εξασφαλίζει όλα αυτά. Στην παρουσίαση λοιπόν αυτής της σύντομης έκθεσης, εγώ έχω γνωμοδότηση, έχω σταθεί σε, στα κυριότερα σημεία και έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι οι συνάδελφοι από τις άλλες πολιτικές ομάδες θα προσθέσουν και άλλα στοιχεία και ήδη εκφράζω τη χαρά μου για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα λάβει η χώρα. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, στα φιλαδικά, κυρία Σάγια. Ο ανταγωνισμός για τις δημόσιες αγορές στην, καλύτερη, στη χειρότερη περίπτωση ε, βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών και μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερη κάλυψη. Υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να βελτιωθεί το καθεστώς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί και η περιβαλλοντική και η κοινωνική πτυχή. Για πολλές επιχειρήσεις ε, πρόκειται για κάτι το οποίο σίγουρα είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά θα, πρέπει να δούμε πώς μπορούν να ληφθούν καλύτερα υπόψη τα στοιχεία αυτά στις ε, κρατικές προμήθειες χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για τις δημόσιες συμβάσεις και να μην απειλείται ο ανταγωνισμός. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ε, όλες μας τις δυνατότητες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, δυνατότητες που μας προσφέρει η παρούσα νομοθεσία, δηλαδή τα στοιχεία μέσω της οποίας δίνεται μια δημόσια σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνουν και κάποια ελάχιστα συγκεκριμένα κριτήρια. Τα ελάχιστα συγκεκριμένα κριτήρια θα μπορούσαν για παράδειγμα να είναι τα στοιχεία που είναι πιο απλά, οι πτυχές της νομοθεσίας ε, στη χή χώρα για παράδειγμα. Στις δημόσιες συμβάσεις γίνονται αποδεκτές επιχειρήσεις που έχουν φυσικά καταβάλει όλες τις ε, κοινωνικές ε, επιδοτήσεις, ε, έχουν πληρώσει τους φόρους και ούτω καθεξής. Αυτά είναι δεδομένα. Αλλά σε πολλές χώρες υπάρχουν και στοιχεία στην ομοθεσία που διασφαλίζουν ότι σε επίπεδο ε, παραγγελίας στις δημόσιες συμβάσεις ε, τηρούνται τα όλα, όλα τα στοιχεία που αφορούν στα κοινωνικές πτυχές. Υπάρχουν για παράδειγμα στη χώρα μου κριτήρια ε, μέσω των οποίων οι υπηρεσίες που ε, διεξάγουν μια κρατική προμήθεια θα πρέπει να τη ε, εξετάζουν κατά πόσον οι επιχειρήσεις τηρούν τις κατάλληλες συνθήκε εργασίας, για παράδειγμα. αυτό που ίσως θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στην έκθεση της εισηγήτριας είναι κατά πόσον μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα κοινωνικά κριτήρια με τον τρόπο που μας τα παρουσιάζει η εισηγήτρια. Σίγουρα είναι σοβαρά στοιχεία, αλλά θα πρέπει ε, να αποτελούν στοιχεία συγκεκριμένη νομοθεσία. Δεν μπορεί να γίνονται σε μια οδηγία ή στο συνοδευτικό ε, κανονισμό μιας οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες γνώσεις πώς γίνονται οι αγορές. Ε, δεν είναι μόνο οι τιμές αυτές οι οποίες έχουν σημασία, αλλά και τα ίδια και τα αγαθά, οι υπηρεσίες που προσφέρονται. Ο τρόπος επιλογής επίσης. αν ε, ο τρόπος επιλογής απομακρύνεται πολύ από τις βασικές πτυχές των δημοσίων συμβάσεων. Δηλαδή, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν επιλέγει, για παράδειγμα, ε, τα καλύτερα στοιχεία που περιλαμβάνει μια πρόταση, αλλά επιλέγει μια επιχείρηση που έχει καλή απόδοση σε θέματα διοξιδίου του άνθρακα ή μείωση των εκπομπών. Σίγουρα πρέπει να ληφθούν και αυτά στοιχεία υπόψη, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε ποιο είναι αυτό που προσφέρει τα καλύτερα αγαθά ή τι καλύτερε υπηρεσίε. Λαμβάνονται βεβαίω υπόψη και οι υπόλοιπε πτυχέ, αλλά πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία. Θα καταθέσω και σχετικώ τροπολογίε. Εδώ τώρα ίσως να υπερβάλλω, ίσως η εισηγήτρια να έχει μάλλον επιθετική προσέγγιση για τις υπεργολαβίες. Οι, οι επιχειρήσεις ε, που αναλαμβάνουν ως υπεργολαβία ένα έργο μπορεί να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ποιοτικέ που δεν μπορούν οι ίδιες να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις λόγω μεγέθους τους. Αλλά Αφού η στιγμή η του αρχή γνωρίζει καλά την αγορά της, θα μπορέσουμε ίσως ε, να μειώσουμε ε, τις απαιτήσει ώστε να διασφαλίζουμε και την πρόσβαση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η εισηγήτρια δεν μπορεί να στιγματίζει συστηματικά όλους τους υπερβολάβους ως κάποιοι που είναι επιχειρήσεις ε, που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ένα τελευταίο στοιχείο οι κοινωνικές υπηρεσίες. Καταρχάς, να πω ότι συμφωνώ με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εισηγήτριας, δηλαδή ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι πολύ ευαίσθητες υπηρεσίες, πρόκειται για υπηρεσίες όπως είναι για παράδειγμα υπηρεσίες φροντίδες σε χρόνιους ασθενείς ε, ή σε ηλικιωμένους ε, επειδή ακριβώ πρόκειται για τέτοιε μορφέ υπηρεσίε μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο να επιβεβαιώσει κάποιο την ποιότητα των υπηρεσιών που προφέρεται αλλά στι κοινωνικέ υπηρεσίε και στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών υπάρχουν πολλέ δυνατότητε να έχουμε υπηρεσίε πολύ καλής ποιότητας όταν επιτρέπουμε τη συμμετοχή σε μικρέ και μισές επιχειρήσει. και σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσουμε να παρέχουμε και θέσει εργασία σε γυναίκε επιχειρηματίε, οι οποίε μπορούν να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και ε, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει λόγος να μην υπάρχουν δημόσιες συμβάσεις για κοινωνικές υπηρεσίες. Υπάρχει τρόπος να γίνονται καλά τα πράγματα, να προσφέρονται υπηρεσίες ποιότητες και να ε, προωθείται το επιχειρηματικό πνεύμα και στον κοινωνικό τομέα και νομίζω ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να καθορίσουμε και τι κριτήρια θα πρέπει να ακολουθούνται και σε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες. Προβλέπω λοιπόν και στη συνεργασία με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ε, κάποιοι άλλοι που ζητούν το λόγο. Η Κομισιόν, υπάρχει εκπρόσωπος. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Ορίστε, στη διάθεσή σας. Καλημέρα σας. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει την Επιτροπή σας για την έκθεση. Την περιμέναμε με ανυπομονησία. Περιμένουμε και το αποτέλεσμα αυτής της τελικής γνωμοδότησης. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας ε, πω κάποια γενικά πράγματα για κάποια σημεία τα οποία κατά την άποψή μας θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη ε, στην ε, μεταρρύθμιση της οδηγίας. Καταρχάς, θα πρέπει να προσέξουμε και να αποφύγουμε αμφίσιμες έννοιες. Διότι αμφίσιμες έννοιες δημιουργούν προβλήματα και στην εφαρμογή των νομοθετικών κειμένων. Ε, η νομική ασάφεια μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και για τις ίδιες επιχειρήσεις αλλά και για τις δημόσιες αρχές και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ο σεβασμός ε, της αρχής της ίσης μεταχείρισης, δηλαδή ε, τη διαφάνεια, την έλλειψη διακρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με αυτή την κοινωνική προσέγγιση στις δημόσιες συμβάσεις, αλλά τα κριτήρια θα πρέπει να καθοριστούν κατά τρόπον ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν με αντικειμενικό τρόπο για να γίνει η κατάλληλη επιλογή των υποψηφίων. Επίσης, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε τη δέουσα ισορροπία μεταξύ ε, της προώθησης των κοινωνικών ε, ε, πτυχών μέσω των δημοσίων συμβάσεων, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να μην δημιουργήσουμε και δυσανάλογο διοικητικό άχθος για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόθεση λοιπόν για των κοινωνικών ε, πτυχών θα πρέπει να γίνει σεβόμενη πλήρως ε, και των ε, κανόνων της εσωτερικής αγοράς, οι οποίοι μας ενδιαφέρουν όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ, κυρία. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω ευχαριστήσω την κυρία για τις παρατηρήσεις της να πω κάτι για την ποιότητα των υπεργολαφικών φορέων. Νομίζω τα ίδια πράγματα πρέπει να ισχύουν για αυτούς τους φορείς όπως και για τους αρχικούς αναδόχους. Υπάρχουν καλές τέτοιες εταιρείες υπεργολαβικές, υπάρχουν και κακές. Αυτό ισχύει για όλες τις εταιρείες. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε τα κριτήρια με τα οποία εμεί θα αποφύγουμε να είναι οι μέτρες και οι κακές εταιρείες οι οποίες παίρνουν αυτές τις συμβάσεις. Σε ό,τι αφορά στην συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων, θα πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα για να μην υφίστανται μια υπερβολική γραφειοκρατική ε, πίεση και υπερφόρτωση εάν τηρούν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα της ε, υγείας και της προστασίας των εργαζομένων και πληρώνουν τους φόρους τους, δεν νομίζω ότι πρέπει να υφίστανται ιδιαίτερη πίεση γραφειοκρατική, θα πρέπει να βρούμε λοιπόν άλλους τρόπους για να καλύψουμε την ε, ε, παροχή, μάλλον την σύναψη συμβάσεων. Μπορούμε να κόβουμε σε κομμάτια να ε, γίνονται οι μεγάλες δημόσιες συμβάσεις σε τμήματα, ώστε τα τμήματα αυτά να είναι προσβάσιμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να είναι να καθορίσουμε τις προϋποθέσεις για μια σύμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφείς και αναγνωρίσιμες αλλά κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να υπάρχει η αρχή ότι για ίσες ε, παροχές θα πρέπει να υπάρχει το ίδιο κόστος και επομένως δεν πρέπει να υπάρξει μια πρόσθετη, ένα πρόσθετο γραφειοκρατικό άχθος. Πίστευα θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει για το θέμα αυτό και είμαι έτοιμη και προσβλέπω στην συμμετοχή των άλλων πολιτικών ομάδων και των σχεδόν συγκεκριτών. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. 12 Ιουνίου είναι η προθεσμία για τι τροπολογίε. Το μεσημέρι θα εξεταστεί η έκθεση αυτή στις 10 Ιουλίου στην Επιτροπή μας. 17 Σεπτεμβρίου το πρωί θα εξεταστούν οι τελικές τροπολογίες και θα ψηφίσουμε την επαύριον ώστε να μπορούμε να δώσουμε γέρος την ε, γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς που αν θέλει ο Θεός και δεν αλλάξει τίποτα θα ψηφίσει στις 10 Οκτωβρίου. Ερχόμαστε στο λουκούμιο σημείο της σημερινής που αφορά το σημείο 26 εκπαίδευση κατάρτιση και Ευρώπη 2020 είναι η γνωμοδόση του κυρίου Λούτβιγ Σον. Όπως είπαμε για την εκπαίδευση, κατάρτιση και την Ευρώπη 2020 είναι μια γνωμοδόση προς την Επιτροπή ε, Πολιτισμού και βλέπω ότι ο κύριος Θέρκας θα αντικαταστήσει τον κύριο Λούντβικ Σον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς ο κύριος Λούντβικ Σον δεν μπόρεσε να είναι εδώ και ζήτησα να σας ενημερώσω εγώ για τις βασικές ε, προτάσεις του προς την Επιτροπή ε, Πολιτισμού για αυτή την πρωτοβουλία. Τέσσερις είναι κατά βάση. Πρώτον, ο κύριος Λούντβιξον υπενθυμίζει στην Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παιδεία και η απόκτηση δεξιοτήτων για να υπάρχει και υψηλό επίπεδο στις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και εν καιρό κρίσης, όχι μόνο για τους ε, νέους, αλλά και για όλο τον παραγωγικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο θέμα το οποίο επισημαίνει, σχετίζεται και με το προηγούμενο βεβαίως, είναι ότι υπάρχει σαφή σχέση μεταξύ του επίπεδου παιδείας και των δυνατοτήτων ε, απασχόλησης που έχουν οι νέοι. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι η παιδεία είναι επένδυση και όχι μόνο δαπάνες. Και όταν φτάνουμε σε ε, σημεία όπως αυτά της δημοσιονομικής ε, πειθαρχία, τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να το θεωρήσουν επένδυση και όχι δαπάνες και όχι να κάνουν περισσότερες περικοπές στην παιδεία όπως δυστυχώς διαπιστώνουμε ακόμα και σε τομέες όπου υπάρχει πολύ περισσότερος κίνδυνος. Για παράδειγμα η ένταξη στον χώρο της εργασίας των νέων. Το τρίτο σημείο που επισημαίνει ο κύριος Λούγκβιξον είναι ότι Κανεί δεν μπορεί να λάβει βοήθεια όταν την έχει ανάγκη αν δεν είναι κατάλληλα ενημερωμένο. Και αυτό φαίνεται ότι ισχύει σε γενικέ γραμμέ, Δηλαδή δεν γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να είναι δικαιούχοι προγραμμάτων ε, τι υπάρχει από πλευρά προγραμμάτων και φυσικά δεν μπορούν να υποφεληθούν αυτών των προγραμμάτων. Και τέλο, ο κύριος Λούτβισον θεωρεί και υπάρχουν πολλέ ενδείξει γι' αυτό ότι το σοβαρότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι και νέες που ε, ολοκληρώνουν ή σταματούν τις σπουδέ τους χωρίς να έχουν λάβει ε, την υποχρεωτική παιδεία που είναι απαραίτητη. Και τι θα πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να μειώσουμε το ποσοστό των ανθρώπων που εγκαταλείπουν ε, τις σπουδέ τους και δεν ολοκληρώνουν την ε, παιδεία τους. Και διότι εδώ, και αυτό το καταδεικνύουν όλα τα στατιστικά στοιχεία, ε, είναι πολύ σημαντική η σχέση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας των ανθρώπων που δεν έχουν περατώσει τις σπουδέ τους ε, και αυτό που είναι πιο σοβαρό είναι ότι ε, αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά αποτελούν το όχημα της παράτυπης εργασίας. Και Υπάρχουν και συγκεκριμένες προθεσμίες. Μέχρι 4 Ιουνίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και θα τις λάβει δε υπόψη ο κύριος Λούτβιχσον. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. κύριο Μπενιόν. Μια δήλωση θέλω να διαβάσω εκ μέρου τη κυρίας Μάνερ, η οποία είναι ο Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι σημαντικά για το μέλλον των νέων ανθρώπων. Πρέπει να βρούμε και σχολεία και δουλειέ για όλου. Η συμβολή τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση μπορεί να μα βοηθήσουν να πετύχουμε του στόχου τη θετική 2020. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να υλοποιηθούν από κάθε κράτο μέλο και οι επενδύσει είναι η απάντηση μακροπρόθεσμα και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Στην παρούσα κρίση πρέπει να βρούμε λύσεις, να προκαλέσουμε ανάπτυξη μέσω των προπολογισμών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, που δυστυχώ δεν είναι βιώσιμη αυτή τη στιγμή. Οι προκλήσει είναι δεδομένε στον τομέα τη αποσχολησιμότητα. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι το κλειδί για την πρόσβαση μεταξύ άλλων και στην ανώτερη εκπαίδευση, για να βελτιώσουμε την κατάσταση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη ανεργία των νέων. Το Εράσμος δίνει νέες δυνατότητες στους ε, νέους να αποκτήσουν εμπειρίες. Έχω υποβάλει τροπολογίες και προσβλέπω σε συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο τον λόγο. Όχι. Η Κομισιόν μήπως εκπροσωπείται. Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί με μια έκθεση πρωτοβουλίας. Και... Κανείς άλλος τον λόγο. Απλώς εγώ θα μεταφέρω όλα αυτά που ελέγχθησα στον κύριο Λούτβιξον. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. 4 Ιουνίου προθεσμία τροπολογιών εξέταση και των συμβαστικών στις 20-21 Ιουνίου και ψηφίζουμε στην Επιτροπή αμέσως μετά για να λάβει υπόψη της το αποτέλεσμα η Επιτροπή Πολιτισμού, Πολιτιστικών Υποθέσεων, στι 10 Ιουλίου. Ολοκληρώσαμε την εξέταση της της διάταξης, δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα, οπότε θα τα ξαναπούμε στις 20 και 21 Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.